για την υλοποίησή του. Βεβαίω, οι χώρε μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την εφαρμογή των δράσεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Λίγη εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στι 12.30. Θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα τη ημερησία διατάξεω, την έκθεση δηλαδή του κυρίου Ντέβα για την υποδομή σε φράγματα στι αναπτυσσόμενε χώρε. Ο κύριο Ντέβα για 4 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σωστά συζητήσαμε εδώ και μισή ώρα, συζητάμε εδώ και μισή ώρα, τις αιτίε και τους τρόπους πρόληψης των περιττών θανάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Η έκθεσή μου για την υποδομή στα φράγματα στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει σαν σκοπό να ασχοληθεί με το ίδιο θέμα, την πρόληψη δηλαδή των περιττών θανάτων από πλημμύρες που προκαλούνται από την υποχώρηση των παγετώνων στο Χιντουκού, στα Χιμαλάια και στη Λατινική Αμερική. <clears throat> Πετώντας ε, στα 18.000 πόδια ε, με ελικόπτερο πάνω από τα Ιμαλάια, είδα κάτι θαυμάσιες υπέροχες ε, λίμνες από κάτω. Και όμως είναι τα πιο επικίνδυνα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. Εν συνεχεία, ε, συναντήθηκα ε, με τους εκπροσώπους του, του Διεθνούς Κέντρου Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης ε, που έχουν εντοπίσει περισσότερο από 8.000 παγετώδεις λίμνες εκ των οποίων 2003 θεωρούνται, 203 ε, συγγνώμη, είναι πολύ επικίνδυνες. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε σεισμούς δεν το αναφέραμε εδώ στην Ευρώπη, αλλά σίγουρα αναφέρθηκε στην Ασία, όπου πέθαναν πολλοί άνθρωποι. Και ήταν 9,69 ε, ε, της κλίμακας Ρίχτερ αυτός ο σεισμός. Ε, με τέτοιες σεισμού σεισμούς μπορεί να ανοίξουν αυτά τα φράγματα. Ο, τρο, λόγος που αυτές οι παγετώδεις λίμνες ε, δημιουργήθηκαν και που είναι φυσικό, φυσικές λίμνες, είναι γιατί οι παγετώνες λιώνουν ε, γρηγορότερα ορισμένες περιόδους του έτους. Το νερό κανονικά από, από αυτούς τους παγετώνες ε, τροφοδοτεί τους μεγαλύτερους ποταμούς, τον Γκάντζι, τον Κίτρινο Ποταμό, τον Τάρι. Τροφοδοτεί λοιπόν αυτές τις ποτάμιες λεκάνες και ε, 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι πίνουν νερό από εκεί και καλλιεργούν ρύζι σε αυτές τις όχθες των ποταμών. Όμως, εξαιτία του επιταχυνόμενου λιωσίματος των παγετώνων και της ισόρεσης αυτού του νερού στις 8.000 παγετώδεις λίμνες που είναι φυσικές, οι οποίες μερικές φορές παθαίνουν ρήξη, έχουμε πλημμύρες και έχουμε τρομακτικές πλημμύρες, όπως συνέβη πρόσφατα στο Πακιστάν, όπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι, 20 εκατομμύρια άνθρωποι, το διανοείστε, έμειναν άστεγοι και χιλιάδες χιλιάδων ανθρώπων πείνασαν. 500.000 άνθρωποι έπρεπε να τους στρέψουμε με επιστηστική βοήθεια και όλη η σοδιά του σιταριού καταστράφηκε για όλο το χρόνο επιστρέφουν ξανά και ξανά οι πλημμύρε. Τον Ιούλιο έγινε ξανά πλημμύρα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μεγάλε εκτάσει ε, του Πακιστάν είναι πλημμυρισμένε. Ακόμα και τη Ινδία. Αυτός ο... Δεν μπορούμε πια να προβλέψουμε τον τρόπο που ε, στέλνει ε, στέλνουν αυτές οι παγετώδεις λίμνες στο νερό σε μεγάλους ποταμούς όπως το Γκάντζι λοιπά, Στο Γιαντζέ. Είναι σημαντικό λοιπόν να επισκευάσουμε αυτές τις λίμνες που δημιουργούνται, που σχηματίζονται με φυσικό τρόπο. Ούτω ώστε να ελέγξουμε του, με κάποια μέτρα μετριασμού του νερού, με συμφώνια, με ανοιχτά κανάλια, με τούνελ, ούτω ώστε να χαμηλώσουμε ε, το επίπεδο νερού σε αυτές τις παγετώδεις λίμνες και να ελέγξουμε το πώς γίνεται στις ποτάμιες λεκάνες και να χρησιμοποιήσουμε το νερό αυτό ε, που υπάρχει εκεί σαν δεξαμενή. Πάρα πολλή δουλειά πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διεθνής υπηρεσία του ΟΗΕ <clears throat> ούτως ώστε η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ, το Μπουτάν και άλλες χώρες να μπορέσουν να συνεργαστούν στα πλαίσια του ΟΗΕ για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Νέβα. Πάμε στην ε, διαδικασία Catch the Eye. Ο πρώτος, και μην ξεχνάτε όλοι ότι έχετε ένα λεπτό, είναι η κυρία Χούμπνερ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, Νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ξέρουμε ότι πολλές χώρες υποφέρουν από καταστροφές εξαιτίας ακατάλληλα κτισμένων φραγμάτων, φραγμάτων που δεν λειτουργούν σωστά ή γιατί δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι με τις κλιματικές αλλαγές που έχουμε τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερες ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες θα συμβαίνουν και θα επαναλαμβάνονται όλο και περισσότερο οι πλημμύρε. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιάξουμε τα καλά τα άλλα συστήματα. Ξέρουμε πώς να τα φτιάξουμε, διότι τα φράγματα δεν απαιτούν νέες κατασκευαστικές τεχνολογίες. Αυτές που χρησιμοποιούν χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν είναι αποτελεσματικές. Θα πρέπει όμως να δώσουμε τεχνογνωσία και εμπειρία να προσφέρουν χώρες αυτές για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Οι πλημμύρες είναι ένα από τα πιο καταστροφικά φυσικά φαινόμενα εξαιτία ε, της απώλειας ανθρώπινων ζώων και του οικονομικού κόστους. Θα πρέπει λοιπόν, ε, λόγω των κλιματικών αλλαγών, να πάρουμε μέτρα, διότι υποφέρουν όλο και περισσότερο οι αναπτυσσόμενε χώρε. Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, διότι οι παγιατόδει λίμνε αποτελούν απειλή. Συμφωνώ με την εισηγητή που λέγει ότι θα υπάρχουν σίγουρα τα μέτρα που θα μπορούν να προλαμβάνουν τέτοιες καταστροφές και ισχυρές βροχοπτώσεις αυξάνουν το κίνδυνο όλο και περισσότερο και μπορεί να σπάσουν τα φράγματα. Βασιζόμενοι στα συμπεράσματα των εμπειρογνωμόνων ξέρουμε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη κάποια πράγματα και γι' αυτό θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνες αυτές τι καταστάσει. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκου. Η, το, το, το νερό παρόλο που καλύπτει 70% του, του πλανήτη είναι στην ουσία σπάνιο αγαθό και επιδεινώνεται η κατάσταση αυτή με τις πλημμύρες και βλέπουμε το παράδοξο Δυστυχώ υπάρχει ένα πρόβλημα με την μετάφραση από τα ρουμανικά. Ελπίζουμε να λυθεί γρήγορα. din cauza reliefului montan sau accidentat. Totodată aceste sisteme... Δυστυχώς δεν υπάρχει μετάφραση από τα ρουμανικά. Dar în cazul în care construcția este defectuoasă... Συνεχίζουμε. Εάν η κατασκευή δεν γίνει ορθά, τότε θα υπάρχουν σημαντικά σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οδήποτε νέα έργα θα πρέπει να βασίζονται πρώτα σε μελέτες, αναλυτικές μελέτες επιπτώσεων που να υπακούν στις αρχές της παγκόσμιας ε, οργάνωσης κατασκευής φραγμάτων. Και αυτό θα πρέπει να το σέβονται όλες οι χώρες. Ευχαριστώ. Δεν μου ζητεί κανείς άλλος ε, να λάβει το λόγο στο, στο σύστημα Eye. Ο Επίτροπος. Κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστώ τον κύριο Ντέβα για την έκθεσή του και που μας ε, εφίστα την προσοχή σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και μας υπενθυμίζει τη σημασία του προβλήματος, που νομίζω ότι επί καιρό ε, δεν ήταν τόσο σοβαρό ή τέλο πάντων δεν ήταν πολύ ψηλά προτεραιότητε τη παγκόσμια τη διεθνού κοινότητα. Ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω εδώ εκ μέρου τη Κομισιόν για να σα μιλήσω για αυτό το θέμα. Θέλω να τονίσω ότι η Κομισιόν συμφωνεί ότι η υποδομή των φραγμάτων ε, έχει μια πολύ, είναι πολυδιάστατη και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ε, ολοκληρωμένο τρόπο. Θα πρέπει να έχουμε μέτρα προσαρμογής, μετριασμού, ε, πολιτικό διάλογο ανάμεσα στις ε, όμορες χώρες επίσης, που είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το ψήφισμα είναι επίκαιρο γιατί εστιάζει σε όλα τα θέματα τα οποία συνδέονται με το χτίσιμα των, χτίσιμο συγγνώμη, των φραγμάτων, την ενίσχυσή τους ε, και την τεχνολογική ε, προσαρμογή τους, ώστε να είναι βιώσιμα και να μειωθούν οι κοινωνικές, πολιτικές και ε, περιβαλλοντικές αρνητικέ επιπτώσεις. Ε, σε διεθνέ επίπεδο, εμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και τι επιπτώσει. Με τι δεσμεύσει στο Κανκούν και στην Κοπενχάγη, η Κομισιόν έχει ε, δεσμευτεί να υποστηρίξει τι αναπτυσσόμενε χώρε να εφαρμόσουν μέτρα προσαρμογή και μετριασμού όπω προλαμβάνονται στην διεθνή αναπτυξιακή στρατηγική και στα σχετικά προγράμματα. Ιδίω σε τοπικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί προγράμματα βιώσιμη ανάπτυξη με μικρέ παρεμβάσει που προσαρμόζονται καλύτερα στο τοπικό περιβάλλον. Επίση, η έκθεση πολύ σωστά τονίζει το, ότι το λιώσιμο των παγετώνων αυξάνει σε όλο τον κόσμο. Και είναι ιδιαίτερα έντονο, όπω πολύ σωστά αναφέρει η έκθεση, στην οροσυρά των Ιμαλαΐων. Το, η επίπτωση είναι ότι έχουμε ε, πολλές επιπτώσεις στις περιοχές κατάντι, ε, σε παραποτάμιες περιοχές και σε έντονα, ε, σε αγροτικές περιοχές. Ιδίως στην Ασία, όπου έχουμε 60.000 παγετώνες και τέτοιες λίμνες. Επομένως, συμφωνούμε ότι οι πλημμύρες που προκαλούνται από την υπερχείληση αυτών των ε, λιμνών πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, και οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διασυνοριακά, να κάνουμε πρόληψη της καταστροφής, να έχουμε προσαρμογή και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Ε, γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε σε επαφή με τοπικά Ινστιτούτα και φορείς, με εμπειρογνώμονες, όπως ε, αυτή η αυτό το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης, καθώς και με κυβερνήσεις των πληττόμενων περιοχών, ούτω ώστε να συζητήσουμε τις δράσεις και τους τρόπους συνεργασίας να υποστηρίξουμε την Ασία ε, στον αγώνα της για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής καθώς και τη διαχείριση ε, των υδάτινων δεξαμινών. Και αυτό περιλαμβάνεται και στις προσπάθειες που θα γίνουν ε, στη συνάντηση που θα γίνει στον Μπουτάν Ευχαριστώ. Πέρα τη συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι η, κυρία, ε, είναι η έκθεση της κυρίας Σίμερ για την ενίσχυση των ε, αναπτυσσομένων χωρών στο να αντιμετωπίσουν